ύπαρξη ενό οικονομικού φορέα που θα μπορεί να απαντήσει σε περίπτωση μη συμμόρφωση ή προβλημάτων που παρουσιάζουν τα ίδια τα προϊόντα. Είναι αδιανόητο πλέον ένα επικίνδυνο προϊόν, πλαστό προϊόν ή που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία να μην ε, έχει κάποιον αρμόδιο. Έχουμε συμπεριλάβει διατάξεις προστασίας των καταναλωτών που αγοράζουν ε, στο διαδίκτυο και οι οποίοι θα πρέπει να απολαύουν την ίδια ασφάλεια όπως ε, με τα προϊόντα που πολλούνται ε, με τον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρεία συνεργασία πολιτική ε, και επιχειρησιακή μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ώστε να υπάρξουν κοινέ στρατηγικέ ε, και να διασφαλίσετε ένα σύστημα ομοιόμορφων και συνεκτικών ελέγχων. Ειδικότερα θέλουμε να εξαλείψουμε το port shopping, όπως ονομάζεται, δηλαδή την ύπαρξη σημείων εισόδου προνομιούχων για τους παραβάτες με μερικές φορές πλήρη απουσία τελωνιακών ελέγχων. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει στόχους ε, και πρότυπα εναρμονισμένα για τους ε, συνοριακούς ελέγχους, κοινέ μεθόδους ε, αξιολογήση κινδύνου, μέγιστο συντονισμό και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των εθνικών αρχών σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού δικτύου. Επιπλέον έχουμε προβλέψει ένα σύστημα επαγρύπνηση όπου δεν θα υπάρχει πλέον περιθώριο για σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου ναι, ούτε ε, προνομιούχος αντιμετώπιση ορισμένων παραβατών. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ε, δημοσίων εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εντείνουν του ελέγχου που θα γίνονται στα κράτη-μέλη βάσει συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ικανοτήτων και προτεραιοτήτων. Επίσης αυξήσαμε τις εξουσίες ε, των εθνικών αρχών, ούτω ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις αποτελεσματικές ε, και στον κόσμο του διαδικτύου όσον αφορά τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα. Αυτά είναι τα βασικότερα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει. Ελπίζω να υπάρξει ευρεία συνένεση επί αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Επιτροπή στο λόγο έχει Επίτροπος κυρία Thank you very much, President. Dear members. Ε, Πρόεδρε, ε, αγαπητοί βουλευτές, χαίρομαι που βλέπω την επιτυχή έκβαση για την επιτυχία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του, αλλά και το σημαντικό αυτό επίτευγμα στη στρατηγική εσωτερικής αγοράς. Ο κανονισμός έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχουμε πάρα πολλά προϊόντα που δεν είναι ασφαλή και που δεν είναι ε, συμμορφωμένα με τις διατάξεις και τα πρότυπα. Έτσι θα έχουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών και πιο δίκαιη εσωτερική ενιαία αγορά για τα προϊόντα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον εισηγητή Νίκολα Ντάντη και ε, τους κοιόδης συγητές ε, Κάρα, Σαλτεμόζο και Ντάλτον. Ήταν τεράστια η προσπάθεια και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει τόσο γρήγορα το θέμα διαφορετικά πριν τις εκλογές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που όλοι μας θα θέλαμε να ήταν διαφορετικά. Πρώτα θα ετοιμάσουμε μια δήλωση για τη νομική βάση. Στη δεύτερη όμως εργαζόμαστε πιο προς μεγαλύτερη ομοιογένεια και ομορφία στους εξωτερικούς ελέγχους, στα εξωτερικά σύνορα, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτής της νομοθεσίας. Θα έχουμε τώρα τη μοναδική ευκαιρία ε, να σταματούμε αυτά τα προϊόντα πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Με ε, αλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών ελεκτικών αρχών και των τελωνιακών αρχών και σε διάφορα άλλα σημεία η πρόταση και θέλω να το τονίσω βελτιώθηκε ακόμα. Εδώ σκέφτομαι ιδιαίτερα ε, τον έλεγχο ομοτήμων Και τώρα πλέον ε, πραγματικά υπάρχει διαφορά ε, και για τους εθνικούς επιθεωρητές. Έχουν οι αρχές καλύτερα εργαλεία και περισσότερες εξουσίες να ελέγχουν προϊόντα που πολλούνται επιγραμμικά και μπορούν οι επιθεωρητές ε, να έρχονται σε επαφή με αυτές τις νέες ψηφιακές μορφές και ψηφιακές αγορές και να τις ελέγχουν καλύτερα και για πολλές κατηγορίες προϊόντων θα έχουμε εκπρόσωπο ε, του κλάδου ή της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι οι αρχές θα μπορούν να απευθύνονται ε, σε εκείνον για να ενημερώνονται καλύτερα για να λύνουν τα προβλήματα συμμόρφωσης. Επίσης, βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών και των επιχειρήσεων ε, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό να προλαμβάνεις τη μη συμμόρφωση παρά να ε, κατάσχεις προϊόντα και να τα απομακρύνεις ε, από την αγορά. Γιατί πολλές επιχειρήσεις ε, είναι καλόπιστες, απλώς δεν γνωρίζουν τι κανόνες ισχύουν για τα προϊόντα. Και στη συνέχεια το τρίτο και ίσως το σημαντικότερο θα βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, τώρα έχουμε πάνω από 500 αρχές επιθεώρησης και ελέγχου της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα ε, κυκλοφορούν απρόσκοπτα εντός των εσωτερικών συνόρων μας. Δυστυχώς η συμμόρφωση και επιβολή του νόμου όχι. Και στις διασυνοριακές ε, περιπτώσεις χρειαζόμαστε εθνικούς επιθεωρητές να συνεργάζονται καλύτερα με τις θελωνιακές αρχές. Θα υπάρξει λοιπόν πανευρωπαϊκή συνεργασία με ένα τέτοιο δίκτυο συμμόρφωση προϊόντων. Ένα στοιχείο λείπει μόνο. Τα χρήματα. Ιδιαίτερα για τη συνεργασία γιατί ο δίκτυο συμμόρφωση που ανέφερα προηγουμένω. τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν από το πρόγραμμα τη εσωτερική αγορά και χαίρομαι πολύ που είχατε ενεργή συμμετοχή και προσήλωση και προσβλέπω και στην περαιτέρω υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό συμβιβασμό με ισορροπία που αντανακλά τις διάφορες απόψεις και τις διάφορες ανησυχίες όλων των ενεχομένων και ελπίζω να το εγκρίνετε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Εκ μέρους Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μικόλασικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η ασφάλεια των καταναλωτών και η προστασία της εσωτερικής αγοράς είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω το σχέδιο κανονισμού που φιλοδοξεί ε, στην διατήρηση και ενίσχυση των εναρμονισμένων κανόνων για ε, τα προϊόντα, όπως είναι παιχνίδια, καθαριστικά, δομικά υλικά, ε, σωρευτές, μπαταρίες, ελαστικά, ζυζανιοκτώνα, ηλεκτρικά απόβλητα και ένα σωρό άλλα προϊόντα. Είναι απαράδεκτο ε, να μπορεί κανείς σήμερα να παρακάμπτει τους ισχύοντες κανόνες. Ακούμε ότι το 32% των παιχνιδιών, 58% των ηλεκτρονικών συσκευών και 47% των δομικών υλικών που ελέγχθηκαν δεν ανταποκρίνονταν στις ε, ε, προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Αυτό είναι θέμα και των ε, καταναλωτών και των εμπόρων. Καλό είναι να έχουμε κέντρα δοκιμών, αλλά καλό είναι να είναι και αξιόπιστες οι μελέτες και οι δοκιμές. Και ε, η πραγματογνωμοσύνη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε τομείς όπως θέλουν ιδιαίτερες γνώσεις, τα επικίνδυνα χημικά που εμφανίζονται σε καλλιτικά και παιχνίδια. Στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει ο κύριος Κάρας για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Ισηγητά, Ντάντι, ε, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη απόπειρα μεταρρύθμισης του συστήματος παρακολούθησης αγοράς ήταν το 2013 και απέτυχε εκτρά. Εδώ και τώρα κάνουμε μια νέα αρχή για το νέο σύστημα παρακολούθησης της αγοράς. Και ήταν επίγουσα ανάγκη και προς το συμφέρον και όφελος των καταναλωτών ανδρών και γυναικών. Γνωρίζουμε ότι κυρίως τα παιχνίδια, τα πυροτεχνήματα ή τα μηχανήματα είναι τα προϊόντα εκείνα ε, που εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα και τα έχουμε διαπιστώσει. Και εμείς φροντίζουμε να αναλαμβάνει την ευθύνη όποιο φέρνει επικίνδυνα εμπορεύματα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Γι' αυτό χρειάζεται να παρακολουθούμε, να επαγρυπνούμε, να επιτηρούμε για να βρίσκουμε εκείνον που φέρνει τα επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά και να ξέρουμε και ποιον θα φέρουμε ενώπιον των ευθυνών του. Θέλουμε να έχουμε και ίδιου κανόνε ε, για όλου. Όλε οι αλλοδαπέ εταιρείε θα πρέπει να τηρούν του ίδιου κανόνε που τηρούν και οι εγχώριε. Ε, χώρες ευρωπαϊκές, δηλαδή στην εσωτερική αγορά, αν θέλουν να δραστηριοποιούνται και εκείνες στην αγορά μας. Μεγάλες εταιρείες, επιγραμμητές, ε, ε, εφοδιαστικές, μέχρι τώρα είχαν εξαίρεση. Τερματίζεται αυτό. Όποιος θεωρεί ότι πρέπει να πουλάει επικίνδυνα προϊόντα, να πληρώνει και το λογαριασμό για να επιστρέφονται τα προϊόντα αυτά και να λαμβάνει την ευθύνη του. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας και παρακαλώ να υποστηριχθεί όσο γίνεται ευρύτερα η έκθεση αυτή. Όπως ήταν αγαστή η συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας Λιστών και Δημοκρατών. Το λόγο έχει η κυρία Σκάλντε Μόζε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει έρθει η ώρα για καλύτερους ελέγχους στις ευρωπαϊκές αγορές. Ω ε, μέλο του Κοινοβουλίου εδώ και 12 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Η καλή είδηση σήμερα λοιπόν είναι ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα ελέγχου και των ε, προϊόντων που πολλούνται ε, online και που προέρχονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια έρευνα στη Δανία έδειξε ότι τα παιχνίδια που αγοράζει κανείς σε online πλατφόρμες παρατηρήθηκε σε ορισμένε πλατφόρμε ότι κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν, με το, δεν συμμορφωνόταν με του κανόνε. Ε, καλό είναι λοιπόν που έχουμε πλέον ε, ε, επιτέλου κανόνε για αυτά τα προϊόντα. Ε, ώστε οι πολίτε μα να μην αγοράζουν επικίνδυνα. και μεταρρυθμιστών, τον λόγο έχει η κυρία Τόμασιτ για ένα λεπτό. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Internet je promijenio način na koji funkcioniramo. Promjene ljudskog ponašanja. To diadiktio άλλαξε to dropo me τον οποίο ζούμε και που συμπεριφερόμαστε. Αυτό είναι προφανές σε όλους τους κλάδους της ζωής. Μεταξύ άλλων ψωνίζουμε διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν πριν το διαδίκτυο. Επειδή το μερίδιο του online εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά. Πολλά πλαστά προϊόντα κυκλοφορούν όλο και περισσότερα και η προστασία των καταναλωτών είναι πλέον δύσκολη. Η συμμόρφωση των προϊόντων θα μειώσει τις περιπτώσεις απάτης και θα ε, ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Και ειδικότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα προϊόντα τρίτων χωρών που συχνά δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να ξεχνάμε την ισορροπία μεταξύ τη προστασία των συμφέροντων και των δικαιωμάτων των πολιτών αφενό και τη διατήρηση των πλέον εκτιμάτων όπω η ταχύτητα, του μειωμένου κόστου και τη απλούστευση του ηλεκτρονικού εμπορίου από την άλλη. Ευχαριστώ. Και δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δύο μήνες αγόρασα ένα νέο σίδερο και πήγα να σιδερώσω και μου κάψε το πουκάμισο. Έχω εδώ ένα συνάδελφο, μια συνάδελφο που έχει τα παιδιά της και τους πήρε παιχνίδια που τραγουδούσαν και δεν μπορούσαν να σταματήσουν να τραγουδάνε. Ξαφνικά με στα μεσάνυχτα άρχισαν να τραγουδάνε και για να σταματήσουν έπρεπε να βγάλεις τις μπαταρίες όλες και να το πετάξεις. Και έχω και ένα τρίτο συνάδελφο που έχει επικίνδυνο πιστολάκι για τα μαλλιά και ε, ε, μπορεί να σου ξεριζώσει τα μαλλιά ή να στα σπρίσει και να πάρεις 20 χρόνια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε τι πουλάνε στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να είναι ασφαλή τα προϊόντα και να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Και έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Διότι εμείς μπορούμε να βελτιώνουμε κάθε μέρα, αν θέλετε, την ε, νομοθεσία του καταναλωτέ. Αλλά αν δεν τηρούνται οι κανόνες, τι να τους κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ. Ενισχύουμε την επιτήρηση και παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι δεν θα τραβήξουν αυτά που τραβάνε σήμερα οι καταναλωτές με τα πιστολάκια ή με κάποιες μπαταρίες ε, ελαττωματικές που εκρήγνεται μέσα στην τσάντα σου. Αυτό το οφείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και πραγματικά ήταν πολύ καλό που το κάνουμε πριν τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε και ο κύκλος των ομιλητών εκ των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο κύριος Σόσνιερτς για ένα λεπτό.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 νέα πρότυπα, κανονισμοί, γραφειοκρατία, περισσότερη έλεγχη, νέες αρχές, πρόστιμα, επιπλοκές, δυσκολίες, περαιτέρω μεγάλα προβλήματα. Όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε σήμερα στην έκθεση για την εποπτεία της αγοράς. Ε, είναι μια ιδέα που μπορεί να μην δουλέψει. Θα πω τα θετικά όμως. Τι θα κάνουμε με την έκθεση αυτή, η οποία να οδηγήσει σε κάτι καλό ε, το οριγκάμι. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, άκουσα τα όσα είπε ο εισηγητής, τα ποσοστά προϊόντων μη ασφαλών. Είναι εντυπωσιακά και ανησυχητικά. Σκεφτείτε το 32% των παιχνιδιών αφορούν τα παιδιά κυρίως το 40% των ε, συστημάτων προστασίας, ε, ατομικής προστασίας. Αφορούν τη δική μας ψυχή, ε, σωματική κυριότητα Αυτά τα ποσοστά με την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους αναπόφευκτα. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες πρόοδοι όπως αυτή που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε εδώ με θετικό αποτέλεσμα, σημαντικό αποτέλεσμα όπως αυτό που συζητάμε. Είναι σημαντική και η ύπαρξη αυτή των οικονομικών φορέων που θα διασφαλίζουν τη συμμορφώση των προϊόντων Θετικά λοιπόν στοιχεία, ωστόσο λυπάμαι. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Στην προηγούμενη θητεία το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ένα πολύ φιλόδοξο κείμενο αφορούσε την ασφάλεια των προϊόντων και αυτό μπλόκαρε στο Συμβούλιο. Ήταν αντίθετη στους, σε κάποιους κανόνες. Κρίμα, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Τέλο πάντων, είμαστε εδώ που είμαστε και τώρα η Επιτροπή που θα έλθει θα πρέπει να το εφαρμόσει σε όλε τι χώρε. Αυτό που θετικά συζητάμε και εγκρίνουμε εδώ και που θα εγκρίνουμε, ελπίζω, αύριο. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί δύο αιτήματα από την κυρία Γραπίνη και τον κύριο Μαριά. Ο Μαριά Μαριάς βλέπω ότι δεν είναι παρόν. Κυρία Γραπίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτός ο κανονισμός έπρεπε να είχε έρθει εδώ και καιρό, διότι Πρέπει να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Αυτά είναι θέματα θεμελιώδη για το μέλλον της Ευρώπης. Και φυσικά χρειάζεται και καλύτερη υποπτία της αγοράς. Γιατί έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πρέπει να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες. Μ' αρέσει η ιδέα και την καλωσορίζω της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου με δείκτε αναφοράς και πρότυπα ελέγχου αλλά ας μην λησμονούμε ότι θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα διεξαγωγής όλων αυτών των ελέγχων στα τελωνία. Επιτόπου, η Τελωνιακή Ένωση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί όπως γνωρίζουμε. Εάν δεν έχουμε αυτό τον κανονισμό και ε, δεν ολοκληρωθεί, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαι πεπισμένη όμως ότι στην επόμενη θητεία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτά τα θέματα. Θα υπερψηφίσω την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζω, Επίτροπε, ο κανονισμός αυτός να μην παραμείνει κενό γράμμα, αλλά να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, το λόγο έχει και πάλι η Επίτροπος κυρία Μπιανκόφσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τη συνεισφορά σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όμως για την προσήλωσή σας και την αφοσίωσή σας στο συγκεκριμένο θέμα. Με την αυριανή σας ψηφοφορία θα εκπέμψετε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για την συμμόρφωση των προϊόντων και την ασφάλειά τους στην εσωτερική αγορά. Είμαι πεπισμένη ότι ο κανονισμός αυτός και η συμφωνία που πετύχαμε ε, είναι και ε, συνολικός και ισόρροπος και όπως σας είπα και προηγουμένως θα εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνιακών αρχών ε, για να προσαρμοστούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Και φυσικά ε, αυτό ε, θα ολοκληρώσει τη δέσμη μέτρων για τα εμπορεύματα και τα αγαθά. Θέλω να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο και τη Ρουμανική Προεδρία για την υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. είμαι πεπισμένη ότι με τον κανονισμό αυτό έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την εσωτερική γνήσια και δίκαιη αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει και πάλι ο συγητής κ. Ντάντη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώντα αυτή την ανταπάντησή μου, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, το ξέχασα στην αρχή, του τους εισηγητέ για τη συνεργασία του για όλου του μήνε ε, όπου εργαστήκαμε σε αυτό το σημαντικό κανονισμό. Ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα και η συνεργασία τη ε, διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου, πρέπει να πω, υπήρξε εξαιρετική. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπιενκόφσκα και την Επιτροπή στις δύσκολες στιγμές ε, όπου χρειαστήκαμε συνεργασία στάθηκαν στο πλάι μας ε, προσπάθησαν να, να διαμεσολαβήσουν για τις δικές μας θέσεις του Συμβούλιο οπότε τους ευχαριστούμε ε, και την Αυστριακή Προεδρία όπου ξεκίνησε αυτή η διαδρομή και τη Ρουμανική Προεδρία όπου τελειώνουν η διαδικασία Ήθελα να πω δύο πράγματα κλείνοντας. Το πρώτο όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, ο κανονισμός αυτός εντάσσεται στο πρόγραμμα Single Market όπου έχουμε εντάξει οικονομικούς πόρους όπως είπε η Επίτροπος που εγγυώνται την ε, δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη θητεία όταν θα καθορίσουμε πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα στην εσωτερική αγορά θα έχουν επικυρωθεί οι πόροι που διαθέτει το Κοινοβούλιο ώστε να έχουμε αυτό που προβλέπουμε στον κανονισμό, μια πρακτικά εφαρμόσιμη επιθεώρηση της αγοράς. Γι' αυτό απαιτούνται πόροι. Ε, κάτι άλλο. Τι θέλουμε να επιτύχουμε με αυτόν τον κανονισμό. Ίση μεταχείριση μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ε, επιχειρήσεων από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ συχνά από τον υπόλοιπο κόσμο επιχειρήσει είχαν ε, ευκολότερη πρόσβαση χωρί να χρειάζεται να συμμορφώνονται τα προϊόντα του με προδιαγραφέ των ευρωπαϊκών αγορών. Εδώ θα έχουμε μια πιο ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ευρωπαϊκών και μη. Το ίδιο ισχύει και για τι διαδικτυακέ επιχειρήσει ε, και για τι επιχειρήσει που λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Τώρα, όσον αφορά την ενιαία αγορά, ε, πρέπει να διασφαλίζουμε ε, την συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους καταναλωτές μας. θα πρέπει να απαιτείται από όλου του οικονομικού φορεί και από όλε τι αρχέ πλήρη σεβασμό των νομοθεσιών και των προτύπων που έχουμε θεσπίσει μέσα στον χρόνο για την προστασία τη ασφαλεία μα και του κοινωνικού μα μοντέλου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στην έκθεση της κυρίας Σάλντε Μόζε με θέμα προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Το λόγο έχει η εισηγήτρια κυρία Σκάλντε Μόζε για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς οι καταναλωτές θα πρέπει πολλά να παραγγέλνουμε επιγραμμικά. Εισιτήρια, παιχνίδια, μουσική και ένα σωρό άλλα. Έχουμε επιλογή ε, επιγραμμικών διαμεσολαβητικών υπηρεσιών και οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν τις ε, υπηρεσίες αυτές που είναι πολλών πάσης φύσεως και η κατάσταση είναι σαν το Far West. Πρέπει ο καθένας να αποδέχεται τους όρους και τις συνθήκες που του προσφέρει, αλλιώς δεν θα έχει παρουσία. Και πολλές από αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αθέμητες συνθήκες χωρίς διαφάνεια. Αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να δημιουργήσουμε νέο χώρο ε, δικαιοσύνης και διαφάνειας για αυτές τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν. Και αυτό προσφέρει ασφάλεια και στους καταναλωτές που αγοράζουν τα προϊόντα. Αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε. Δεν πετύχαμε όλα όσα επιθυμούσαμε, όμως πετύχαμε μια αρχή. Δημιουργήσαμε ένα θεμέλιο για την νομοθεσία που θα εξασφαλίσει καλύτερη ρύθμιση της επιγραμμικής αγοράς με τη δημιουργία πολύ, πολύ μεγαλύτερης διαφάνειας και ζήτηση για μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, είναι καταπληκτικό. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο καταφέραμε να επιτύχουμε είναι όταν χρησιμοποιεί κανείς επιγραμμικές υπηρεσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ε, πρέπει να είναι πολύ πιο δίκαιες. Έχει διαμακρόν συζητηθεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση αυτή, γιατί έτσι υπάρχει καλύτερη δικαιοσύνη. Οι επιχειρήσεις ξέρουν σε τι εμπλέκονται όταν ζητούν μια τέτοια υπηρεσία. Πετύχαμε πολλά. Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει όριο 15 ημερών για την, ε, για τη λήξη των όρων. Εμείς είπαμε ότι θα μπορεί αυτό να ακυρωθεί αν οι κανόνες δεν είναι παρκώς θετικοί και επιβάλαμε ε, συνθήκες διαφάνειας σε πολλές περιπτώσεις όπως παραδείγματο χάρη οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των, της κάθε πλατφόρμας είναι σαφής. Πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι προποθέσει που με βάση τις οποίες ταξινομούνται. Αυτό είναι σημαντικό επίσης θέσαμε το θέμα της περίοδου προειδοποίησης κατά τη, όταν πρόκειται για λήξη σύμβασης και επίσης μελετήσαμε τις μηχανές αναζήτησης και υπογραμμίσαμε τη σημασία των κανόνων που ισχύουν σχετικά. Όταν οι κανόνες εφαρμόζονται αυτό θα γίνεται, πρέπει να γίνεται με τάξη. Εξασφαλίσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται σωστά, ιδάλλως δεν θα υπάρχει προστασία. Περνάμε λοιπόν σε ένα νομοθέτημα για το χώρο αυτό και θα πρέπει σύντομα να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Εξού και ε, θεσπίσαμε ένα μακρύ μακροσκελή κατάλογο απαιτήσεων του τι πρέπει να αναθεωρηθεί όταν θα αξιολογηθεί και πάλι το νομοθέτημα. Κυρίως όμως πρέπει να πούμε ότι το θετικό εδώ είναι ότι δημιουργείται περισσότερη διαφάνεια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ε, τέτοιου είδους επιγραμμικές ενδιάμεσες υπηρεσίες και μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ισοτιμία για τις επιχειρήσεις στο επιγραμμικό κόσμο και αυτό θα επηρεάσει και τους καταναλωτές που αγοράζουν ε, ε, από τις πλατφόρμες Αυτέ αγαθά και υπηρεσίε. Το να παίρνει κανεί αυτό για το οποίο, το οποίο πληρώνει είναι πολύ σημαντικό. Και εμεί θέτουμε παγκόσμια πρότυπα για τις πλατφόρμες αυτές. Είναι σημαντική ημέρα αυτή. Θέλω να βοηθήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Ευχαριστώ. Των νομικών θεμάτων, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι έχω τη χαρά να μιλώ εξ ονόματος Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε πολύ στενά, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ακούσαμε, οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αναθέτουν σε πλατφόρμες, ακόμα και μικρές επιχειρήσεις, ε, για να φτάνουν στους καταναλωτές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ε, πιο δίκαιο και πιο διαφανές. Στη Μάλτα είχα και εγώ επαφές και συζητήσεις για το θέμα και ε, με ρωτούν τι, μας, κάνει η Ευρώπη για να μας βοηθήσει να προαγούμε τον τουρισμό μας. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού θέλουν περισσότερες πληροφορίες και ε, Επίσης, αυτό που θέλουμε είναι μια ε, μετάβαση στην ψηφιακή ε, οικονομία, στην καινοτομία και σε ένα πιο δίκαιο ε, επιχειρηματικό περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο δίκαιη επιλογή για τους καταναλωτές και όχι μόνο ότι προτείνουν μεγάλες εταιρείες. Το της Επιτροπής, το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Γκάμπριελ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την εισηγήτρια την κυρία Σάλντε Μόζε και τους κοιόδης εισηγήτες για όλες τις προσπάθειές σας, το επικοδομητικό σας πνεύμα, πνεύμα συνεργασίας για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα τόσο γρήγορα. Το Κοινοβούλιο ενίσχυσε το κείμενο, το βελτίωσε ε, οι τροπολογία σας θα βοηθήσουν να υπάρξει ένα περιβάλλον πιο δίκαιο ε, για τις επιχειρήσεις στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Αυτό θα είναι και προς όφελος των καταναλωτών ε, με ένα σύνολο κανόνων σαφές και ένα κανονιστικό πλαίσιο πιο προβλέψιμο. Αυτό με τη σειρά του θα έρθει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο διασυνοριακό εμπόριο. Και έτσι οι πλατφόρμες θα αναπτυχθούν, θα επενδύσουν και θα καινοτομήσουν. Ε, μερικά από τα στοιχεία που πρότεινε το Κοινοβούλιο θα βοηθήσουν πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω αυτών των πλατφορμών να φτάσουν στους πελάτες τους. Το Κοινοβούλιο κάλυψε ένα έλλειμμα ε, στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ε, δεν νοείται να ε, εκφεύγουν των ευθυνών τους και χαίρομαι και για ε, την συγγραφή υποχρεώσεων που προτείνεται έτσι ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση ε, ανάμεσα ε, στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τους πελάτες τους και στην κατάργηση κάποιων πρακτικών. Αυτό λοιπόν το νέο εργαλείο θα είναι ισχυρό, αυτός ο κανονισμός και θα συνεισφέρει στο βασικό μας στόχο που είναι η αύξηση της διαφάνειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό ζήτημα της ταξινόμησης. Παράδειγμα, ακούστηκε προηγουμένως, το είπε η συγγήτρια, εκτός από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οι μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες για ποιο λόγο έχουν διακριτική μεταχείριση στις πλατφόρμες. Επιχειρήσεις ε, Επομένως, ε, το εξή θα μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα το θέμα των διενέξεων και των διαφορών. Θα πρέπει όλες οι πλατφόρμες να έχουν ένα εσωτερικό σύστημα διαμεσολάβησης και εκ των προτέρων να λέγουν ποιος είναι ο διαμεσολαβητής για να υπάρχει εξοδικαστικό συμβιβασμός και διακανονισμός των διαφορών. Ε, αυτό λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των εταιριών. Το τελικό κείμενο ενισχύει και το ρόλο των κρατών μελών στην υλοποίηση και ε, εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για να εφαρμόζονται σωστά οι νέοι κανόνες και αποτελεσματικά. Επίσης, θα πρέπει να συνεργάζονται μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθούν τους νέους κανόνες, να τους αξιολογούν και να μοιράζονται μαζί μας ε, τις ε, πληροφορίες. Δεν σταματά εδώ η δουλειά όμω, Έχουμε χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για περισσότερη σαφήνεια για τον τρόπο λειτουργία των πλατφορμών και των μηχανών αναζήτησης ε, ω προ την ταξινόμησή τους. Θα συνεργαστούμε με τον κλάδο για κανόνες διοντολογία που θα έρθουν να συμπληρώσουν ε, τους κανόνες. Χαίρομαι που διαφυλάζεται η προσέγγιση και το πνεύμα της αρχικής μας πρότασης χάνεται μια σωστή ισορροπία και επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες να αναπτυχθούν. Είναι μια πρώτη μόνο κίνηση αυτή, θα ακολουθήσουν κι άλλες και θυμίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που αυτό τον καιρό εκπονούν μια προσωρινή έκθεση. Ε, θα κατατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Θα προωθήσουμε και θα προχωρήσουμε βέβαια και με την αναθεώρηση όπως προβλέπει ο κανονισμός. 1,5 ε, χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ υπάρχει αυστηρή αναθεώρηση, αξιολόγηση και προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη για να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ελπίζω επίσης το Κοινοβούλιο αύριο να εγκρίνει τον κανονισμό στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, το λόγο έχει η κυρία Ζάμπορσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, οι διαδικτυακές πλατφόρμες αποτελούν μια καταπληκτική ευκαιρία για οικογενειακές επιχειρήσεις, ε, startup, ε, μικρά Airbnb, μικρές επιχειρήσεις, ε, να ξεκινήσουν δραστηριότητες, να απασχολήσουν ανθρώπους και να παρέχουν υπηρεσίες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για αυτές τις επιχειρήσεις. Ο συμβιβασμός που έχουμε επιτύχει μπορεί να ε, είναι ευρύτερο από ό,τι είχα θελήσει εγώ στην αρχή. Στην γνωμοδότησή μου στην Ήτρε είχα προσπαθήσει να περιορίσω τη ρυθμίση στο ελάχιστο. Δεν μπορούμε εμεί να επιβάλλουμε, πιστεύω, επιχειρηματικά μοντέλα. Απλά να καθιερώνουμε ένα σαφέ νομικό πλαίσιο παρόλα αυτά. Μπορώ να υποστηρίξω τη συμβαστική πρόταση με ήσυχη τη συνείδησή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου που υποστήριξαν τη δική μου προσέγγιση στην Ήτρε και θα ήθελα να συγχαρώ επίση την κυρία Σάλντε Μόνσε και τον κύριο Σουφάτο και ο Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει ο κύριο Ζιβέν για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, από τα μεταγάλα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φυσικά η ενιαία αγορά. Παρά τα ελαττώματα του, προτιμώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη χώρα μου να πουλούν σε όλους τους Ευρωπαίους τα 500 εκατομμύρια παρά μόνο στους Γάλλους. Και σήμερα κάνουμε άλλο ένα βήμα, δημιουργούμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Σε αυτή τη νέα ψηφιακή οικονομία που δεν έχει κανόνε, εμεί εξοπλίζουμε την Ένωση με του δικού τη κανόνε, ώστε να μην υφιστάμεθα ξένε νομοθεσίε ούτε τον νόμο των ισχυρότερων οικονομιών. Ειδικότερα εμποδίζουμε στις πλατφόρμες πλέον να επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και οι σχέσεις μεταξύ των πλατφορμών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να, γίνουν, να είναι πιο ισορροπημένες. Φυσικά το εθνικό δίκαιο ε, θα ήταν ανεπαρκέ όταν κλείνει ένας Γάλλος ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία μέσω μια πλατφόρμα που βρίσκεται στην Ιρλανδία ποιο εθνικό δίκαιο ισχύει το γαλλικό, το ιταλικό, το ιρλανδικό Όπω καταλαβαίνετε, δεν λειτουργεί έτσι η κατάσταση. Χρειάζονται ευρωπαϊκοί κανόνε. Και αυτό κάνουμε εδώ. Προστατεύουμε τι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και να τι προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα πρέπει να του προσφέρουμε προστασία μέσω ενό ευρωπαϊκού εναρμονισμένου και κοινού δικαίου για τα 27 κράτη-μέλη. Στο κείμενο αυτό το Κοινοβούλιο έδειξε ότι αποτελεί ένα δημοκρατικό εργαλείο που δεν υπακούει σε λόμπι ούτε σε συμφέροντα. Εγώ είχα την τιμή να είμαι εδώ μέλο για δύο θητείε και κύριε Πρόεδρε, τη στιγμή που εγκαταλείπω το Κοινοβούλιο πλέον, δεν έχω παρά να πω ένα πράγμα. Κρατήστε το ζωντανό. Σα ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει αντιπρόεδρο κυρία Γκέπχαρτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σάλτερ Μόλζα και να τη συγχαρώ για την εξαιρετική της δουλειά. Και εξ ονόματος της ομάδας μας, σοσιαλιστές και δημοκράτες, πρέπει να πούμε ότι ε, είμαστε απολύτως στο πλευρό της και συνιστούμε υπερψήφιση αύριο. Το Booking, το Apple Store, e-dreams, πλατφόρμες που σήμερα ε, παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο έχουν μερίδιο αγοράς και εξουσία στην αγορά. Ε, αλλά αυτό συμβαδίζει με μειωμένα δικαιώματα των χρηστών. Ο σημερινός κανονισμός ε, φέρνει δικαιοσύνη στις πλατφόρμες με απαιτήσει διαφάνειας, με απαγόρευση αθέμητων εμπορικών πρακτικών, με βελτίωση της διαμεσολάβησης και ε, με πιο αποτελεσματική επιβολή του δικαίου. Αλλά και με ένα ειδικό παρατηρητήριο για τις πλατφόρμες, τις επιγραμμικές, ε, γίνεται η εποπτεία καλύτερη και αποτελεσματικότερη. Όλα αυτά είναι καλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές, άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Χαράντσοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κλειδί για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η ειλικρίνεια, η διαφάνεια με τους πελάτες αλλά και με τους εταίρους. Αυτός ο κανονισμός διασφαλίζει αυτή τη διαφάνεια που είναι τόσο αναγκαία χωρίς να επιβάλλει υπερβολικές ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες και τους εμπόρους. Το online εμπόριο είναι το μέλλον της οικονομίας μας. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μια λάθος προσέγγιση να ικανοποιήσουμε τους διεθνείς εταίρους. Κύριε Πρόεδρε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ορισμένοι εδώ θεώρησαν τον κανονισμό ως πολιτικό εργαλείο που θα αλλάξει την πολιτική ανταγωνισμού με, από την πίσω πόρτα. Χαίρομαι που τελικά επικράτησε η κοινή λογική και δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια που έδειξε θάρρος, κατάφερε να επιτύχει μια καλή ισορροπημένη συμφωνία αντί να καταλήξει σε μια που θα επηρεάζει αρνητικά την οικονομία μας και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα του Άλντε θα υποστηρίξει την έκβαση του τριλόγου αύριο στην ψηφοφορία και ενθαρρύνω και τόσο τις πλατφόρμες όσο και τους εμπόρους να χρησιμοποιούν αυτή τη νέα διαφάνεια και να την αξιοποιούν στο μέγιστο. Μόνο υιοθετώντα βέλτιστες πρακτικές και επαρκή ρύθμιση αυτή η αγορά θα είναι δίκαιη για όλους. Φοβάμαι ότι αν οι πλατφόρμες δεν χρησιμοποιήσουν ε, αυτή την ευκαιρία δεν θα έχουν δεύτερη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει η κυρία Ρέντα για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν οι πλατφόρμες είναι σπουδαία ευκαιρία για τις μικρές ευρωπαϊκές εταιρείες. Είτε είναι κάποιος ε, που αναπτύσσει λογισμικό ή πουλάει τα προϊόντα του, οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους μικρούς παίκτες να ανταγωνίζονται τους μεγάλους και να φτάνουν σε πελάτες που ποτέ δεν θα έφταναν διαφορετικά. Αυτό καμιά φορά είναι ο λόγος που κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ήθελαν να αναβληθεί αυτός ο κανονισμός, μάλλον να επεκταθεί ε, με τρόπο όχι λογικό. Οι μεγάλες πλατφόρμες όμως μπορούν να υπαγορεύουν αθέμητες πρακτικές στους πελάτες. Ο δικός μας κανονισμός φέρνει και δικαιοσύνη και διαφάνεια στην αγορά αυτή και αυτό πραγματικά ε, είναι χάρη στο σταθερό χέρι της εισηγήτριας Σάλντε που δεν αφήνει ασίδωτες τις πλατφόρμες, αλλά να μην υπάρχουν και υπερβολικές απαιτήσει που θα σήμαινε το θάνατο του εμποράκου στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εκείνους που συνεισέφεραν ε, προς τη δουλειά αυτή και χαίρομαι που υπάρχει τέτοια μεγάλη συνένεση για τις πλατφόρμες. Σας ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντάντι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Γκάμπριελ, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κανονισμό αυτό ε, επανισορροπεί τι οικονομικέ σχέσει μεταξύ των μεγάλων πλατφορμών και ενό εκατομμυρίου και πάνω ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσω online διαμεσολαβητών και εξαρτώνται από αυτού. Με του νέου κανόνε θα έχουμε καλύτερη διαφάνεια για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε που παρέχονται online περισσότερη ενημέρωση για τις παραμέτρους που καθορίζουν τη θέση μιας προσφοράς ε, στην ιστοσελίδα, ε, υπεράσπιση από μονομερείς ε, αλλαγές όρων και προϋποθέσεων συμβάσεων από τις πλατφόρμες. Οι κανόνες αυτοί θα είναι εποφελείς λοιπόν για εκατομμύρια πολίτες που πολύ συχνά επιλέγουν να αγοράσουν online για καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη επιλογή και ποικιλία και έτσι θα ενημερώνονται καλύτερα. Σε αυτούς τους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι δεν κάμπτεται μπροστά στα συμφέροντα των ψηφιακών γιγάντων, αλλά ότι προστατεύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γράφοντας νέους κανόνες που θα προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το μειονεκ... τη μειονεκτούσα πλευρά ε, των συμβάσεων. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα για τη διαδικασία του Catch the Eye, επομένω το λόγο εξ ονόματο τη Επιτροπής έχει η επίτροπο κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα για μια φορά να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους. Θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά. Ω Επιτροπή χαιρόμαστε για τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον κανονισμό αυτών. Όπως είπατε πολύ σωστά, ε, ε, ε, αποτυπώνει μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών απόψεων και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων. Μια θετική ψήφο λοιπόν για αυτόν τον κανονισμό θα στείλει ένα σαφέ μήνυμα προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει του και του Ευρωπαίου πολίτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να διαφυλάξει την διαφάνεια και την προβλεψιμότητα στι online πλατφόρμες. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε κυρία Σαλντεμός, κυρία Εισηγήτρια και ευχαριστώ και όλους όσοι συνέβαλαν στην ταχεία διεκπαιρέωση του θέματος αυτού. Χαρί στην κοινή μας συνεργασία κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ε, το λόγο έχει η συγκήτρια κυρία Σκάλτε Μόζε για δύο λεπτά. Øh, Ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Χαίρομαι πολύ που πετύχαμε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα θέτει παράδειγμα για τις επιχειρήσεις και για τις πλατφόρμες. Είμαι βεβαία ότι θα ωφεληθούν και οι καταναλωτές μας. Αν δεν είχαμε συνεργαστεί τόσο καλά, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τόσο καλό. Ευχαριστώ λοιπόν στη Ρουμανική, τη Ρουμανική Προεδρία. Είχαμε σκληρές αλλά καλές διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι είχαμε επιτυχία. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ την Κομισιόν και την Επίτροπο. Αν δεν είχατε συμμετάσχει εσείς, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαστε ανοιχτοί σε συνεισφορά και συνεργασία όταν πραγματικά συμβαίνει αυτό, θέλουμε να κάνουμε, επιτυγχάνουμε πολλά για τους καταναλωτές και έχουμε ένα ε, αποτέλεσμα που μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένα πρώτο βήμα βεβαίως και προσβλέπω στη συνέχιση της δουλειάς για να δούμε τι θα προκύψει από το παρατηρητήριο και με το νομοθέτημα αυτό μπορούμε πιστεύω να στείλουμε ένα σήμα από την Ευρώπη προς τον κόσμο για το τι χρειάζεται για αυτό το είδους του κανονισμού, τη διαφάνεια και την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Έληξε η ψηφοφορία, θα κεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στην έκθεση του κυρίου Ντάλτον με θέμα καλύτερη επιβολή και εξυγχρονισμός των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά ο εισηγητής κυρίος Ντάλτον. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πακέτο φέρνει το θέμα των, των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην Επιτροπή του Διαδικτύου. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, ε, τη Ρουμανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους για την επίτευξη συμφωνίας πρώτων ευρωεκλογών. Είχαμε τρεις εβδομάδες από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Επικεντρωθήκαμε σε ένα θέμα ε, μετά από μια πολύ μακριά ημέρα, 10 ώρες διαπραγματεύσεων, καταλήξαμε σε συμφωνία Όπω Όπως πολλοί θα γνωρίζετε, η συμφωνία αυτή υπέστη περαιτέρω διόρθωση από την Κομισιόν και κατέστη σαφέ ε, στη συζητήση ότι έπρεπε να επιβεβαιωθεί η εντολή τη. Έτσι λοιπόν το τελευταίο, το τελικό κείμενο ε, άλλαξε λίγο, αλλά η ουσία παραμένει. Δεν μπορεί κανεί να παραπλανηθεί ω καταναλωτή από προϊόντα που ε, ε, ε, τίθενται σε εμπορία στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Με την συμφωνία αύριο θα σταματήσει αυτή η κατάξη εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι πολλοί πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα και έχουν υποβληθεί τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση για αύριο. Αλλά θα είμαι σαφή. Αν εγκριθεί οποιαδήποτε από αυτέ τι τροπολογίε, θα καταρρεύσει ολόκληρη συμφωνία. Το, το Συμβούλιο και η Κομισιόν κατέστησαν σαφέ ότι έχουν φτάσει στα όρια του, δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Αν λοιπόν περάσουν τροπολογίε, δεν θα υπάρχει υπάρξει συμφωνία. Καμία, ε, ε, καμία ε, ε, διάταξη για την διπλή ποιότητα πριν τι ευρωεκλογέ. Αυτό δεν θα βοηθήσει του καταναλωτέ που αυτή τη στιγμή παραπλανώνται, δεν θα υπάρξει νομοθέτημα υπέρ αυτών. Δεν θα βοηθηθούν οι αρχέ προστασία των καταναλωτών. Δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα για την επιβολή των άλλων ε, διατάξεων και δεν θα, ε, θα ε, συνεχίσει η υπονόμευση των διαφόρων επιχειρήσεων από άλλους. Θα υπάρξουν καθυστέρηση των προσπαθειών για την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος επί χρόνια. Αλλά με αυτή τη συμφωνία πετύχαμε μια αναρχή. Η διπλή ποιότητα αντιμετωπίζεται και θα πρέπει να δει το θέμα με σοβαρότητα η Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, ουσία και όχι μη ρεαλιστικές τροπολογίες. Και το πακέτο αυτό δεν αφορά μόνο τη διπλή ποιότητα. Γίνεται σοβαρή προστασία των καταναλωτών. Και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου καλύφθηκαν σε πολλούς τομείς. Έχουμε, ας πούμε, ε, μια αλλαγή με βάση έναν ε, νέο νόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας ε, καλλιτέχνης δεν θα αναγκαστεί να να, κάποιος δεν θα μπορεί να, να πληρώνει την ίδια τιμή πολλές φορές γιατί αυτό αποτελεί απάτη. Επίσης βάλαμε ε, απαιτήσει για την ε, εμπιστοσύνη και επίσης την ε, ταξινόμηση και την μείωση της τιμής. Όλα αυτά προς όφελος του καταναλωτή. Στην εποχή του διαδικτύου θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τον ενημερωμένο καταναλωτή. Το διαδίκτυο περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες που δίνουν ουσία στον καταναλωτή, αλλά πρέπει να είναι αληθινές. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή σημαίνει ότι αυτοί θα γνωρίζουν όταν λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες. Χαίρομαι που μπορέσαμε να πάρουμε την υποστήριξη της Επιτροπής και του Συμβουλίου για να χτίσουμε την ε, ε, γνώση του καταναλωτή για τα δικαιώματά του. Το ECR, η, μια εφαρμογή που θα αφορά τους καταναλωτές που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, θα τους δώσει ε, άμεση πρόσβαση στην διαδικασία υποβολής παραπώνων που θα λύνουν τα προβλήματά τους. Επίσης, το θέμα της υπαναχώρησης έχει, έχει αντιμετωπιστεί. Αν μπορούμε αύριο να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή, θα έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από την θέσπιση της πρότασης την Επιτροπή, την έγκριση της πρόταση τη Επιτροπής μέχρι την έγκριση. Σας ευχαριστώ όλους, τη Γραμματεία επίσης, τη Νομική Υπηρεσία για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή του. Οι κανόνες αυτοί θα κάνουν πραγματικά ε, σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα του καταναλωτή και α μην καθυστερήσουμε ούτε καν μια μέρα, α εγκρίνουμε το κείμενο αύριο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, το λόγο έχει η κυρία Πέρα Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάλτον και του συνεισηγητέ, του κοιόδη και την Επιτροπή ΜΚΟ. Έκαναν σκληρή δουλειά ώστε να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα είναι καλύτερο από την πρόταση της Κομισιόν σε πολλά θέματα και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που επέμεινε τόσο πολύ στη βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές. Επιπλέον όμως η οδηγία αυτή θα ενισχύσει την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών με πιο εναρμονισμένες κυρώσεις με τις αρχές καταναλωτών ε, σε όλα τα κράτη-μέλη που θα μπορούν να ε, επιβάλλουν πρόστιμα σε εταιρείε με πάνω από 4% του κύκλου εργασιών τους σε περίπτωση ε, βλάβη στους καταναλωτές. Ε, όσοι έχουν υποστεί βλάβη θα μπορούν να ζητούν ε, καταγγελία συμβάσεων ή αποζημιώσεις. Αυτό θα διευκολύνει και τις δικαστικές και εξοδικαστικές διαφορές. Η οδηγία εισάγει διάφορα νέα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση online των καταναλωτών και να βελτιώνεται η διαφάνεια online. Απαγορεύουμε την εμφάνιση ε, ψεύτικων ε, κριτικών από πελάτες. Θέλουμε προβολή των χορηγών ε, στους διάφορους τόπους αγορών. Δεν θα υπάρχουν πλέον ψεύτικες εκπτώσεις για κάποια προϊόντα που θα παραπλανούν τους καταναλωτές και θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ακόμα και αν έχει συμφωνήσει σε, μια, σε ένα συμβόλαιο ένας καταναλωτής ε, ε, έχει δικαιώματα. Όσον αφορά το θέμα της ποιότητας, πολλοί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ε, το μάχονται κατά αυτού εδώ και χρόνια. Αυτό βοήθησε στο να εστιαστεί η προσοχή περισσότερο στο ζήτημα αυτό και να συμπεριληφθεί το ζήτημα στην πολιτική ατζέντα. Έτσι λοιπόν είμαι περήφανη που η Επιτροπή στη Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές για πρώτη φορά πρότεινε νομοθετική νομοθέτημα για το ζήτημα αυτό, ώστε η διπλή μεταχείριση των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει και ώστε ο νέος κανόνας να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα αυτό υπήρξε ευαίσθητο κατά τις διαπραγματεύσεις και το κείμενο που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι συμβιβαστική πρόταση που επιτεύχθηκε από τις διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μετά από και συμφωνώ με τον κύριο Ντάλτο πολύ σκληρέ διαπραγματεύσει, αλλά θα έλεγα επικοδομητικέ. Θέλουμε ο ιδιωτικό τομέα να αναλάβει ευθύνε και να σταματήσει τη διπλή ποιότητα. Τώρα είναι απολύτω σαφέ. Δεν μπορούν να κλέβουν σε θέματα ποιότητα και να πουλούν με την ίδια συσκευασία προϊόντα με σημαντικά διαφορετική σύνθεση. Αυτό είναι σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Χαίρομαι που ήδη τώρα υπό την πίεση που ασκήσαμε πολλοί κατασκευαστές προσάρμοσαν τις συνθέσεις των προϊόντων εναρμονίζοντα τις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περαιτέρω βήματα που κάναμε με την Omnibus πρόταση και για την online ανταλλαγή. Ε, ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις ε, εξαλείφουν τις διαφορές ε, και με τις μόνιμες δοκιμές που κάνουμε τώρα είδαμε ότι υπήρχαν πολλά προϊόντα παραπλανητικά στην αγορά που τώρα θα εξαφανιστούν. Ε, ελπίζω τώρα θα σταματήσει αυτή η διαφεροποίηση από τους παραγωγούς και όσοι συνεχίσουν θα πρέπει να την αιτιολογούν. Οι έμποροι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται, θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να αποδεικνύουν ε, για ποιο λόγο αιτιολογούν τέτοια διαφορά. Οπότε το blacklisting, ε, η συμπερίληψη σε μαύρη λίστα οποιασδήποτε τέτοια πρακτική θεωρούμε ότι δεν είναι καλή λύση. Ο μηχανισμός ε, του αθέμητου εμπορίου θεσπίζεται στο άρθρο 6 και όχι στη κατάρτιση μαύρης λίστας. Το άρθρο 6 είναι αποτελεσματικό. Το άρθρο 6 του UCPD χρησιμοποιείται διαρκώ ω νομική βάση από τις Εθνικές Αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο πρόσφατα, για παράδειγμα, οι Ιταλικές Αρχές το χρησιμοποίησαν για να επιβάλλουν πρόστιμο στη Wizard και στην Ryanair για την παραπλάνηση ε, των καταναλωτών όσον αφορά την πραγματική τιμή των εισιτηρίων τους. Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών στα κράτη-μέλη βασίζουν πολλές από τις υποθέσεις του σε αυτό το άρθρο. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ε, το αποτέλεσμα μια δράση κατά πέντε εταιριών ενικές αυτοκινήτων, επειδή δεν ήταν σαφή όσον αφορά το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρήχαν ε, με ανεπαρκή ενημέρωση. Και έτσι θα εξακολουθήσει η ε, κατάσταση και στο μέλλον όσον αφορά την παράνομη χρήση διπλή ποιότητα. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτού του νομοθετήματο και θα συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ε, εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Φέτο πάλι προτείνουμε ένα εκατομμύριο ευρώ χορηγίε ε, από το πρόγραμμα για τους καταναλωτές για αυτό το θέμα και χάρη σε ένα πιλωτικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δεσμεύσουμε ένα 660 ε, εκατομμύρια, 1.200.000 χορηγίες ε, στις ε, ενός καταναλωτών για καλύτερες δοκιμές. Μετά έχουμε μια ρήτρα αναθεώρηση στο κείμενο, σαφή. Δεσμευόμαστε να επαρεξετάσουμε την κατάσταση δύο χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, ώστε να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να καταστήσουμε τις λύσεις πιο αυστηρές. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ελπίδα ότι η οδηγία αυτή θα εξυγχρονίσει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 Η οδηγία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, προσφέρει πράγματι καλέ λύσει στου καταναλωτές, αλλά δεν ε, αντιμετωπίζει το ουσιαστικό πρόβλημα, δηλαδή την διαφορετική ποιότητα των προϊόντων που ε, ε, παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει ένας κατάλογος των δικαιολογημένων εξαιρέσεων, όπως είπε η Κομισιόν. Δικαιολογημένες εξαιρέσει. Αυτό σημαίνει ότι η οδηγία δεν απαγορεύει ουσιαστικά τι αθέμητε πρακτικέ. Εγώ πήγα στο Κίλ στη Γερμανία και αγόρασα τυρί κρεμόδες τυρί που λέει ότι είναι, έχει γάλα 100% ενώ στην Κρακοβία περιλαμβάνει, περιλαμβάνει σκόνη γάλακτος. Επίσης ένα τυρί Φιλαδέλφια το οποίο ε, ε, Αγόρασα τσάι στην Κρακοβία και έχει 1% από ξηραμένα φρούτα και 50 φορές περισσότερη ποσότητα στο ίδιο τσάι που αγόρασα στο Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν εγώ και άλλοι 100 συνάδελφοι υπογράψαμε μια τροπολογία που ...παγορεύει άνευ όρων αυτή την πρακτική. Θέλω την υποστήριξή σας, γιατί δεν υπάρχουν καλοί και κακοί καταναλωτές στην Ευρώπη. Η ίση αγορά πρέπει να είναι ίση για... την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει για δύο λεπτά η Αντιπρόεδρος κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά πρέπει να πω ότι σε αυτό το πακέτο μέτρο που έχουμε να ψηφίσουμε αύριο έχουμε πάρα πολλές καλές προτάσεις και τεράστιες βελτιώσεις για τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, για τους καταναλωτές, άνδρες και γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, αλλά και την Επίτροπο και την Προεδρία του Συμβουλίου, που εργάστηκαν άοκνα. Σε αυτά τα θετικά μέτρα είναι ο εξυγχρονισμός των πλατφορμών. Εκεί έχουμε συμπεριλάβει και τέτοιες υπηρεσίες που αμείβονται και με δεδομένα. Κάποιες πλατφόρμες που υποτίθεται ότι είναι δωρεάν, δεν είναι δωρεάν, τις πληρώνουμε με τα δεδομένα μας. Θα πρέπει να υπάρχει και νομική ε, αρρωγή για τους πολίτες, ε, τους καταναλωτές και κάτι άλλο που μέχρι τώρα δεν υπήρχε σε αυτό το τομέα, κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόστιμα που είναι τουλάχιστον 4% του ετησίου κύκλου εργασιών της